Η Τουρκία είναι μια χώρα υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να υπάρχουν διαπραγματεύσει και πρόοδο πρέπει να υπάρχει αμοιβαία πρόοδο. Θέλουμε να λάβουμε το θέμα της Τουρκίας στα σοβαρά, οπότε είναι απαραίτητο να τονίσουμε πότε υπάρχουν πρόοδοι, αλλά όταν υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Αυτά τα γεγονότα σε σχέση με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία δεν είναι καινούρια. Εμείς με μεγάλη έκπληξη είδαμε τις ε, ε, συλλήψεις εναντίον δημοσιογράφων και εναντίον μέσων ενημέρωσης στο παρελθόν με την ευκαιρία των διαδηλώσεων στο Γκεζί Πάρκ και χθε είδαμε να επαναλαμβάνονται τέτοιες ενέργειες και νιώθουμε βαθιά ανησυχία γιατί με τον τρόπο αυτό διακόπτεται ο πρόεδρος Entwicklung ε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι γίνονται αυτές οι ενέργειες κατά των μέσων ενημέρωσης αντιπολίτευσης. Πρέπει να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση για όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε την οδό της ε, αντιπαράθεσης και των αντιπίνων κατά των δημοσιογράφων που δεν έχουν την ίδια άποψη με μας. Ζήτησα λοιπόν αμέσως από την τουρκική πρεσβεία να μας δώσει εξηγήσεις και διευκρινήσεις για τα θέματα αυτά και εξ ονόματός σας λέω ότι θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή αλλά και μεγάλη ανησυχία τα τεκτενόμενα στην Τουρκία.